της συνεδρίασης θα υποβληθούν προ έγκριση την επόμενη φορά και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει. Ε, τα ψηφίσματα που μόλις εγκρίναμε θα τα διαβιβάσουμε στους ε, αποδέκτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνει εδώ μια